Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open the meeting of Committee Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Ρέτζη σήμερα το απόγευμα. Είμαστε λίγοι ακόμα, αλλά είμαι πεπισμένη ότι θα προσέλθουν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, και ευτυχώ έχουν έρθει και κάποιοι άντρε ε, γιατί στην αρχή θεώρησα ότι θα πρέπει να πω μόνο αγαπητέ συνάδελφοι. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με την έγκριση του σχεδίου της σα διάταξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια σε σχέση με την ημερήσια διάταξη τη σημερινή συνεδρίασης. Εάν όχι, θεωρούμε το σχέδιο της σα διάταξη ω συγκεκριμένο. Το επόμενο σημείο είναι ανακοινώσει τη Προέδρου. Έχω μια σειρά από ανακοινώσει να σα κάνω σήμερα, ενημερωτικού χαρακτήρα. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από κοινού με τον κύριο Βανίστελνο και τον Λουίς Βέστιβαλ στις 8 και 9 Ιουνίου παρευρέθηκα σε ένα άτυπο συμβούλιο ε, των Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχή στη Βαλέτα, που διοργανώθηκε βέβαια από την ε, Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου. Το κύριο λοιπόν θέμα ήταν η αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους ε, πολίτες σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία αλλά και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής. Είχαμε μάλιστα τη δυνατότητα να ακούσουμε τις θέσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής ε, και εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ εδώ σήμερα είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν τη μελλοντική περαιτέρω ανάπτυξη της ε, πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο τώρα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές αν θέλετε απόψεων και υπάρχουν κάποιες ομάδες κατ' μελών. Μία ομάδα υποστηρίζει τη μελλοντική ευελιξία της πολιτικής συνοχής και τις δυνατότητες, ε, και την ύπαρξη δυνατοτήτων ε, να αντιδρούμε στα τεκτενόμενα σε καθημερινή βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως για παράδειγμα δηλαδή στο ζήτημα της μετανάστευσης, την προσφυγική κρίση και ούτω καθεξής. Από εκεί και μετά υπάρχει μια άλλη ομάδα κρατών μελών που υποστηρίζουν περισσότερο τη διατήρηση ε, της ε, πολιτικής συνοχής με τον ε, τρόπο που αυτή είναι διαμορφωμένη σήμερα. Άλλες, μια άλλη πρόκληση για τα κράτη-μέλη είναι ε, η δυνατότητα ε, διαφοροποίησης ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής μεταξύ των κρατών μελών, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις διαδικασίες ελέγχου, σε ό,τι αφορά γενικότερα τη δυνατότητα του να προσαρμόζεται καλύτερα η πολιτική στις ανάγκες, στις κάστοτε ανάγκες των κρατών μελών. Αυτά ήταν επιμέρου ζητήματα, αλλά το κυρίως μήνυμα είναι ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειές τους χρειάζονται την ε, πολιτική συνοχή. Αντιλαμβανόμαστε τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να επιτείνουμε τι προσπάθειε μα έτσι ώστε τα αποτελέσματα τη πολιτική συνοχή να είναι πιο απτά, πιο ορατά, πιο αντιληπτά από του πολιτέ μα. Δηλαδή θα πρέπει να του δώσουμε να καταλάβουν ποια είναι αυτά τα επιτεύγματα τη ε, πολιτική συνοχή. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια αποτελέσματα της, ε, του άτυπου συμβουλίου στην Μάλτα η δική μας ε, παρουσίαση από την πλευρά του Κοινοβουλίου έγινε αμέσως μετά από τον και όπως είχε αναφέρει και η έκθεσή μας ε, η αρθρωτή των ε, Building Blocks, ε, αναφέραμε και συγκεκριμένα ποιοι είναι οι δικοί μας στόχοι σε σχέση με την μελλοντική πολιτική συνοχή. Και θα πρέπει να πω ότι ορισμένε αντιπροσωπείε, εθνικέ δηλαδή των κρατών μελών, είχαν πραγματικά εντυπωσιαστεί από το ενδιαφέρον που δείχνουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου για το μέλλον της πολιτική συνοχή. Δεύτερη τώρα ανακοίνωση από την πλευρά μου αφορά στην ε, έκτακτη συνεδρίαση της, των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και μάλιστα έτσι σε κάποιο άτυπο περιβάλλον γιατί συναντηθήκαμε σε ένα όμορφο σατό και όχι εδώ στις ε, Βρυξέλλες. Παρ' όλα αυτά βέβαια δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε αν θέλετε λίγο ε, το περιβάλλον εκεί γιατί είχαμε πολύ εντατικές συζητήσεις με τρία κυρίως ε, θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν το Brexit ε, όπου ο κύριος Μπαρνιέ μας έκανε μια γενική παρουσίαση των ε, προετοιμασιών των προπαρασκευαστικών εργασιών για τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ξεκινήσαν ε, σήμερα, όπως γνωρίζετε. Και όλοι οι πρόεδροι των Επιτροπών ανταποκρίθηκαν στα όσα μας παρουσίασε, λέγοντας ότι αντιλαμβανόμαστε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία οι διαπραγματεύσεις θα θέλετε, θα ακολουθήσουν δύο διαφορετικά στάδια. Αλλά ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει κάθε μία από τις επιτροπές να αναλάβει το δικό της ρόλο στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων με βάση δηλαδή και τους τομείς ε, πολιτική που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, έτσι ώστε να εμπλακούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως επιτροπές σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πάντως ο κύριο ε, Βαν ε, και ο κύριο ε, Χώσταρ, αλλά και ο πρόεδρος Ταγιάννη, είπαν ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από το ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών δηλαδή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως επίκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει το πρώτο θέμα προς διαπραγμάτευση. Το δεύτερο θα είναι η ε, χρηματική αποσημείωση. Ε, αυτό βέβαια είναι ένα ιδιαίτερο, ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα, αλλά εάν δεν βρεθούν λύσεις, δεν ληφθούν αποφάσεις σε σχέση με αυτά τα δύο κύρια ζητήματα, δεν θα είναι δυνατόν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε σχέση με τα πιο λεπτομερή άλλα, δηλαδή ζητήματα προς διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η κύρια θέση που θέλει να υιοθετήσει ο κύριος ε, Μπανιέ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν σήμερα. Και σε αυτή του την τοποθέτηση υποστηρίζεται πλήρω από τον κύριο Βερχόφστατ. Το δεύτερο τώρα ζήτημα που συζητήσαμε ήταν η συμφωνία σε συνεργασίες ε, με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά ε, ζητήματα και νομοθετικά και μη νομοθετικά ή θέματα ε, νομοθετικά και μη νομοθετικά, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον διορισμό των αρμοδίων επιτροπών από την πλευρά του Κοινοβουλίου και την σύγκρουση, αν θέλετε, εδώ που μπορεί να υπάρχει σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε, αλλά και τον κανόνα 55 και τον κανόνα δηλαδή των συναρμόδιων επιτροπών. Η δική μας τώρα η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, βρίσκεται κάπου στη μέση, αν θέλετε. Γιατί σε άλλες επιτροπές υπάρχουν πάρα πολλά ε, αντικρουόμενα ε, συμφέροντα ε, σε σχέση με άλλες επιτροπές. Εμείς δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει τέτοια σύγκρουση συμφερόντων με άλλες επιτροπές και εγώ εξέφρασα την τοποθέτηση της Επιτροπής Ρέτζη ότι δηλαδή θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αρμοδιότητε που έχουμε σήμερα, αλλά προφανώ είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με άλλε επιτροπέ, εφόσον με αυτόν τον τρόπο ε, συνεργαζόμαστε αποτελεσματικότερα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη σύνταξη εκθέσεων. Ε, και εδώ αναφέρθηκα σε κάποια, ε, για παράδειγμα στην έκθεση Νοβάκοβ, συνεργασία δηλαδή με την Επιτροπή Προπολογισμών. Αλλά και άλλε συνεργασίε που έχουμε επιτέχει με άλλε επιτροπέ. Οπότε Αυτά ήταν τα δύο κυρίως ζητήματα που συζητήσαμε στο πλαίσιο της ενόγκος συνεδρίασης και υπήρξε στο τέλος και ένα δείπνο όπου πήρε το λόγο ο πρόεδρος Σταγιάννη και ο οποίος τόνισε την ανάγκη πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πολίτες μας σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις πολιτικές της Ένωσης και αναφέρθηκε στην διακήρυξη της Ρώμης ε, κατά τον εορτασμό της εξωτερικής της Ένωσης. Αυτά ήταν τα κυρίω ε, συστήματα που ανέφερε ο κ. Σταγιάννη. Αυτά λοιπόν ήταν οι ανακοινώσει από την πλευρά μου σε ό,τι αφορά τα όσα έγιναν κατά τι τελευταίε ημέρε. Από εδώ και πέρα, ε, να σας πω ότι για το μέλλον έχουμε έναν ε, πολύ φορτωμένο μήνα. Έχουμε 26 και 27 Ιουνίου θα υπάρξει μια αρκετά μεγάλη από, ε, ε, αντιπροσωπεία ουσιαστικά από την Επιτροπή μας ε, στο φόρουμ όπου εγώ μαζί με την κυρία Κρέλ και την κυρία Βέρσφαλ θα πάρω το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής μας και όπου θα αναλάβω και ως συντονίστρια ενό από τα πάνελ συζήτηση. Από εκεί και μετά θα υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση το πρωί της 29ης Ιουνίου ε, ε, σε σχέση με μια κοινή ακρόαση σε ό,τι αφορά την ατζέντα για τις ε, πόλεις, urban agenda και εδώ η γραμματεία θα σας αποστείλει και την ημερήσια διάταξη το ταχύτερο δυνατό και μετά 12 και 13 Ιουλίου θα λάβει χώρα η επόμενη τακτική μας συνεδρίαση όπου θα προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων με την πούμε την Εστονική δηλαδή Προεδρία του Συμβουλίου, όπως και το Επίτροπο Βεστάγκερ σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσει. Και, και με Επίτροπο Κρέτσο, οπότε δύο Επιτρόπους. σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ε, δυνητικές μελλοντικές εργασίε τη Επιτροπή, σε ό,τι αφορά το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Θα σταματήσω πάντως εδώ με τις ανακοινώσεις μου, γιατί ήταν αρκετές ε, για σήμερα και επειδή έχουμε α, πολύ φορτωμένη ημέρα σε διαταξή σήμερα, οπότε θα συνεχίσουμε με τις εργασίες μας. Ε, έχουμε λοιπόν το workshop το οποίο οργανώνεται από το τμήμα σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή και την κλιματική αλλαγή. Ζητήθηκε αρκετά. Αρχικά το workshop από την δική μας επιτροπή με τίτλο «Την εξέταση ε, του ρόλου της ε, πολιτικής συνοχής» ε, και είχαμε εδώ συντάξει και μία έκθεση πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά την ρόλο που μπορούν να παίξουν οι πολίτες στην εφαρμογή των στόχων της Συμφωνίας των Παρισιών COP21. Και ε, έχουμε την κυρία Βαλινό σε σχέση με αυτήν την έκθεση από την πλευρά μα. Ε, έχετε λοιπόν μπροστά σα εδώ το, την ημερήσια διάταξη στο πρόγραμμα του workshop και οι ομιλητές μας θα αναφερθούν ε, σε διάφορα ζητήματα όπως τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών παγκόσμιων θεματολογίων, τον ρόλο της πολιτικής στις πόλεις και πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σχετικών στόχων. Ξεκινάμε λοιπόν, περνάμε τώρα στην μέση διάταξη του workshop και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρτιν Νέσμπιτ, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, του προγράμματος ε, διακυβέρνησης ε, κλίματος και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Πολιτική. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Νέσμπιτ για την πολιτική συνοχή και τους στόχους της Συμφωνία των Παρισιών. Έχετε το λόγο κύριε Νέσμπιτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή σας που μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να σας παρουσιάσω το έργο μας. Θα περιγράψω το περιεχόμενο της εκθεσής μας, η οποία υπάρχει και εδώ στην είσοδο. Και θα αρχίσω λέγοντας ότι κοιτάξαμε ποια είναι η εμπειρία που έχουμε από την προηγούμενη περίοδο συνοχής την προηγούμενη περίοδο πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου που ήταν ε, μέχρι το 2014, 2007-2014. Μετά θα δούμε τι γίνεται στην σημερινή προγραμματική περίοδο 2014 με 2020. Τι μαθήματα έχουμε πάρει από την εμπειρία μας αυτή και πώς αξιολογούμε και τις επιπτώσεις της Συμφωνίας των Παρισίων. Στη συνέχεια περιγράφουμε και κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να γίνει μετά το 2020, την επόμενη περίοδο πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Εισαγωγικά δεν θα σας εκπλήξουν αυτά ότι έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την κλιματική αλλαγή υπάρχει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, υπάρχει το πρωτόκολλο του Κιώτο και υπάρχει βέβαια και η Συμφωνία των Παρισίων που λέει ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 2 βαθμούς, 1,5 ουσιαστικά, τονίζοντας ιδιαίτερα το ρόλο που μπορούν να παίξουν σε αυτό οι πόλεις και οι διάφορες τοπικές αρχές που καλούνται να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους, τις δράσεις τους και να ανταλλάξουν πρακτικές μεταξύ τους. Υπάρχει τώρα το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το πακέτο 2020, τι προβλέπουμε για το 2020, τι θέλουμε να πετύχουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας κλιματικά για το 2020, να μειωθούν κατά 20% οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, 20% επίσης ε, να παίρνουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και βελτίωση επίσης κατά 20% στην απόδοση. Όλα αυτά ε, σίγουρα συνεισφέρουν πολύ το τι, έχει γίνει, τι θα έχει γίνει δηλαδή μέχρι το 2020 για το πώς θα προγραμματίσουμε τη συνέχεια. Ε, αντίστοιχα και για το 2030. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δούμε και ποια είναι η αστική διάσταση. Το θέμα της υπαίθρου είναι κάτι το οποίο θα θίξω αργότερα. Ποιε είναι οι εμπειρίε που έχουμε τώρα από την πολιτική συνοχή στην περίοδο 2007-2013. Η κλιματική δράση Νομίζω ότι για πολλούς ήταν ένας νέος τομέας ε, επενδύσεων. Με ενεργειακή απόδοση, για παράδειγμα. Και σίγουρα ήταν μια δύσκολη πορεία εκμάθησης αυτή. Διαπιστώσαμε επίσης ότι πολλές φορές δεν υπήρχε καλά διαρθρωμένη καλά διαρθρωμένος τρόπος για να αξιολογήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα για τον καθορισμό των στόχων. Ο καθένα μόνος του έβαζε τους στόχου του και προσπαθούσε να βρει πώς θα τους πετύχαινε. Έπειτα το θέμα τη σχέση ε, κόστους και αποτελεσματικότητας. Δεν ήταν πάντα ότι καλύτερο, δεν ήταν πάντα προτεραιότητα. Και τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης ε, δείχνουν διάφορα γενικά συστήματα στο δημόσιο τομέα. Γενικότερα για αυτό το θέμα ήταν σαφές ότι υπήρχαν επιπτώσεις στον προγραμματισμό των χωρών μελών που είχαν σαν αποτέλεσμα οι συνομοθέτες να αποφασίσουν πιο συγκεκριμένους στόχους για την ενεργειακή αυτή απόδοση. Και μερικές φορές οι περιφέρειες ε, χρησιμοποιούσαν επιχορηγήσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. κυρίως για την επιχορήγηση νοικοκυριών χαμηλών εσόδων. Δεν έφτανε όμως αυτό, οπότε τελικά επιδοτήθηκαν δάνεια για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα νοικοκυριά από το Ταμείο Συνοχής. Είχαμε κάποιες πρώτες εμπειρίες με τα χρηματοδοτικά μέσα, νέα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το Τζέσικα ακριβώς για την ε, ενεργειακή απόδοση. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα δεν υπήρξε συνολική ε, σχεδιασμένη δομή για τις επιπτώσεις των επενδύσεών μας για το κλίμα. Έρχομαι τώρα στην περίοδο 2014-2020. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε δέσμευση τουλάχιστον 20% από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό να πηγαίνει ε, σε θέματα που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και την περιορίζουν. Θέλαμε βελτίωση της συνοχής και της ακρίβειας. Όντως υπήρξε βελτίωση στη διαδικασία, στην επικοινωνία, όπως δείχνουν οι διάφοροι δείκτες. Όμως, είναι ακόμα δύσκολο να καθορίσουμε το ακριβές επίπεδο της συμβολής της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Κάποιες, ε, κάποια βοήθεια σίγουρα υπήρξε όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου, αλλά δεν έχουμε συνολικά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στι δαπάνες, ε, χρησιμοποίησαμε διάφορα μέσα, τη συμφωνία εταιρική σχέση, την εξάντε ερεσιμότητα και διάφορους θεματικού στόχου σχετικού με το κλίμα. Ο ένα, για παράδειγμα, είναι ο τέσσερα που αναφέρεται στην οικονομία χαμηλού άνθρακα και ο πέντε, στόχος 5, που έχει να κάνει με την αδοχή ε, του κλίματος. Πώς δηλαδή θα περιοριστεί η κλιματική αλλαγή. Και υπάρχει και ο έξι ο οποίος αποτελεί μια γενικότερη περιβαλλοντική κατηγορία και στην πράξη απορροφά πολλές επενδύσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Τώρα πρέπει εδώ να σας προειδοποιήσω ότι αυτό είναι κάτι που το έχω προσθέσει, δεν το έχετε στα χαρτιά τα οποία σας μοίρασα. Και εδώ περιγράφουμε πώς ε, έγινε ε, η οικονομική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Με τη βοήθεια σε ένα μεγάλο βαθμό. Πρέπει να ξέρουμε ότι το κλίμα είναι ένας βασικός ε, στόχος 100%. Είναι στόχος της δαπάνης, αλλά τελικά το 40% πήγε εκεί. Συνεπώς, για την πολιτική συνοχή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ο μηχανισμός εκείνος ο οποίος βοήθησε περισσότερο σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όμως χρησιμοποιούνται και πιο συγκεκριμένοι κώδικες 133 στον αριθμό, πιο συγκεκριμένοι ε, κώδικες για την αξιολόγηση των δαπανών των επενδύσεων που έγιναν σε σχέση με το κλίμα. Αυτούς τους κώδικες θα τους βρείτε στο παράρτημα αριθμός 1. Αλλά εδώ στη διαφάνεια αυτή έχω βάλει κάποια παραδείγματα για την ενέργεια, 100% για ποδηλατόδρομους επίσης και επίσης οι δαπάνες για λιμάνια που το θέμα της διαχείρισης των υδάτων μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής επίσης. Βάσει των κωδικών λοιπόν έχουμε καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα. Όπως είπα, είναι ε, ο μηχανισμός ο πιο περίπλοκος αλλά και ο πιο έγκυρος που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Σίγουρα όμως το να έχει κανείς ένα κωδικό για κάθε επένδυση απλοποιεί κάπως ε, την εικόνα. Μερικές φορές ε, υποτιμούμε τις επενδύσεις, μερικές φορές τις υπερτιμούμε. Και περνώ στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ εμφανίζεται το τμήμα στήριξης για κλιματικές δράσεις βάση του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου, μάλλον των διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων. Βλέπετε εδώ για την κάθε χώρα, βλέπετε και το μεσόωρο 5,1%. Πάντως δεν πρέπει τα στοιχεία αυτά να τα πάρετε 100% για την Αυστρία, ας πούμε. Νομίζω ότι έχουν συμπεριληφθεί πάρα πολλές δαπάνες και βάσει άλλων ε, κανονισμών. Οπότε είμαστε πολύ ε, σκεπτικοί κατά πόσο η γενοδορία αυτή που αντικατοπτρίζεται σε αυτή τη διαφάνεια όσον αφορά την Αυστρία είναι πραγματικότητα ή όχι. Τώρα για τους θεματικούς στόχους πάλι. Εδώ βλέπετε ότι οι κυριότερες επενδύσεις των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για το κλίμα επάνε στους στόχους 4, 5 και 6 που είναι για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Επίσης όσον αφορά την αντίσταση στην κλιματική αλλαγή. Αλλά, όπως είπα και νωρίτερα, πολύ μεγάλη συνεισφορά πάει στον θεματικό στόχο 6 που είναι υπέρ του περιβάλλοντος, προστασία του περιβάλλοντος. Στην επόμενη διαφάνεια συνοψίζονται οι δαπάνες, από πού προέρχονται. Και εδώ βασιζόμαστε σε, ως πηγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της του 2016. Και εδώ φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συνεισφέρει σημαντικά. Το Ταμείο Συνοχής επίσης, η συνοχή συνεισφέρει κατά πολύ στους περιβαλλοντικούς στόχους, κάτι το οποίο μπορεί να εκπλήξει κάποιους. Όπως θα γνωρίζετε επίσης, η πολιτική συνοχής έχει μια πολύ σημαντική διάσταση που αφορά τις πόλεις και την εδαφική συνεργασία. Υπάρχουν λοιπόν συνεργασίες ανάμεσα στην κλιματική δράση και άλλες δράσεις, τις οποίες θα αναφερθούν σίγουρα άλλοι ομιλητές αργότερα. Αλλά σύντομα θέλω να αναφερθώ στην ενεργειακή απόδοση. Οι επενδύσεις στον τομέα αυτών είναι πολύ σημαντικές για την εντόπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης στρατηγικές για να έχουμε χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Και εδώ παίζει ρόλο η κινητικότητα. Και έρχομαι και στο τρίτο που είναι η αναζωγόνηση, η αναγέννηση και η απορρίπανση βιομηχανικών χώρων. Η συμφωνία του Παρισιού φυσικά ενισχύει τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, την ανάγκη δηλαδή να έχουμε αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει, ε, πιο φιλόδοξες ε, δράσεις επίσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και θα λέγαμε επίσης ότι απαιτεί πολιτικές και επενδύσεις τώρα για μακροπρόθεσμα σχέδια προκειμένου να καταργηθεί ο άνθρακας σαν πηγή ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τώρα να γίνει αυτό για να μπει η Ευρώπη στο σωστό δρόμο και να μην χρησιμοποιεί πλέον άνθρακα το 2040 ή 2050. Το άλλο που λέμε για μετά το 2020 είναι ότι επειδή μηδέν οι αρνητικές ακόμα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα χρειάζονταν από τις βιομηχανοποιημένες χώρες για να πετύχουμε τους στόχους, κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό επικεντρωνόμαστε πολύ και στην χρήση γης. και θέλουμε σε αυτό να βοηθήσει και το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης Εδώ φυσικά επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην Ήπεθρο και μας ενδιαφέρει η διαχείριση των αποβλήτων και η αστικοποίηση όταν γίνεται να γίνεται αποτελεσματικά και αποδοτικά. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των στόχων της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής και της συνοχής. Και φυσικά να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας κλίμα σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις δράσεις. Επίσης πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τη Συμφωνία των Παρισίων. Και έτσι καταλήγουμε στα εξή συμπεράσματα. Παρόλο που η συμπερίληψη του κλίματος όλες μας τις δράσεις για την περίοδο 14 με 20 αποτελεί ένα βήμα προς τα μπρος, χρειάζονται περισσότερες αλλαγές μετά το 2020 και κυρίως να δούμε τα προγράμματα συνοχής και οι στόχοι, οι άμβλες των επιπτώσεων ε, στο περιβάλλον, πώς θα προχωρήσουν. Επίσης, η αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων του Παρισιού να γίνονται με, πιο, με τρόπο πιο στάνταρτ, από όλους δηλαδή με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, σύμφωνα και με την πρωτοβουλία της Επιτροπής Budget Focused on Results, προπολογισμό δηλαδή που να κρίνεται βάσει των αποτελεσμάτων, και εμείς θέλουμε να δούμε τι θα έχουμε ως αποτέλεσμα από την συνεισφορά της μελλοντικής συνοχής όσον αφορά τις δαπάνες που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Συμφωνία των Παρισίων είναι βέβαια πολύ απαιτητική, αλλά πιστεύουμε εφικτή. Όπως είπα και νωρίτερα, απαιτεί περισσότερη συνεισφορά από όλου και συμβατότητα με τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν να κάνουν με την απαλλαγή από τον άνθρακα. Πρέπει να αποφεύγονται λοιπόν επενδύσεις όπου το αποτέλεσμα είναι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να λάβουμε υπόψη μας και τις εξάντε ερεσιμότητες και όλα όσα έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα με την παρουσίαση του κυρίου Ραφαήλ Τούτς σχέσεις δηλαδή μεταξύ στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, συμφωνίας Παρισιού και νέας νεοαστικού θεματολογίου. Είναι διευθύνση προγράμματος στο Union Habitat το κύριο Τας παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που προσκαλέσατε τον ΟΗΕ. Είμαστε μια υπηρεσία του ΟΗΕ υπεύθυνη για τις πόλεις και τις αστικές περιοχές. επόμενα δέκα λεπτά θα ήθελα να σας μιλήσω για την σχέση μεταξύ Συμφωνίας Παρισιού και νέου αστικού θεματολογίου που υιοθέτησαν πέρσι στο Κίτο όλες χώρες του ΙΕ. Να σας δείξω ακριβώς πώς σχετίζονται αυτές οι δύο ατζέντες, τα δύο θεματολόγια και παρουσιάσουμε κάποια συμπεράσματα. Πράγματι, Αυτά τα τρία θεματολόγια για την κλιματική αλλαγή σχετίζονται στενά. Να δούμε το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα δούμε πάνω από το ίμιση των στόχων αφορούν άμεσα τους ΟΤΑ, την τοπική διακυβέρνηση. Δηλαδή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ελοπιθούν χωρίς την πλήρη υποστήριξη των ΟΤΑ. Στη Συμφωνία των Παρισιών, από τους 160 συμμετέχοντες, το 69% μιλούσαν για αστικά μέτρα και στο αστικό θεματολόγιο 22% των αφορών αφορούν την κλιματική αλλαγή κατά μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο την προηγούμενη απόφαση που αφορούσε το Habitat τα αντιτήματα όπου είχαν πολύ χαμηλότερο ποσοστό βλέπετε λοιπόν ότι σχετίζονται άμεσα και αλληλοεξαρτώνται αυτά ο ρόλος των πόλεων τώρα ιδιαίτερα όσον αφορά την κλιματική συμφωνία έχει γίνει όλο και πιο σημαντικός από το 2007 και η συμφωνία του Παρισιού αναφέρει ξεκάθαρα τις υποεθνικές αρχές ως ε, συμβαλόμενα μέρη, ενώ παλαιότερα είχαμε μόνο αναφορά στην κοινωνία των πολιτών και τους ζητάει η συμφωνία να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να μοιραστούν και να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα για την οποία θα μοιράζονται οι πολίτες. Λίγα παραδείγματα. Και αυτά είναι παραδείγματα που είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο αρχικά όσον αφορά τον μετριασμό της αμβλήσης. Καταρχάς τι μεταφορές, αστικές μεταφορές που είναι ένας τομέα κλειδί σημαντικών επιτυχιών. Μιλάμε εδώ συγκεκριμένα για βιώσιμα συστήματα μεταφορών για όλους. Στο νέο αστικό θεματολόγιο υπάρχει μια ιδιαίτερη έμφαση όσον αφορά συστήματα αποδοτικά όσον αφορά τους πόρους, συστήματα μεταφορών. Και ξέρουμε ότι στο παρελθόν όλες οι πόλεις είχαν αναλάβει δράση με σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την μείωση των εκπομπών, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Όσλο. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και με άλλα κομμάτια του πλανήτη, όπως η Ινδονησία που συνεργάζονται με την Ένωση, με την ΔΕΦΚΟ και λαμβάνουν χρηματοδότηση και ιδιαίτερα η πόλη του Μπογκόρ στην Ινδονησία για την ανάπτυξη ταχύων συστημάτων μεταφορών, για τη μείωση βεβαίω τη εξωτερική συμφόρηση αλλά και των ρήπων. Παρόμοια θα μπορούσαμε να πούμε και για τον τομέα των κτηρίων, που για αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, τομέα όσον αφορά την άμβληση. Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε δύο στόχους συγκεκριμένα που λαμβάνουν υπόψη μας για την άμβληση και βέβαια αυτό αφορά και τον Βορρά και τον Νότο, αφορά και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και τις πρωτοβουλίες τους και εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα από την Κοπεχάνη και το Παρίσι όπου τα κτίρια πραγματικά διαπρέπουν στην ε, μείωση των εκπομπών. Όπως σας έλεγα συμβαίνει και στο Νότο Ήδη υποστηρίξαμε αφρικανικές χώρες για την ανάπτυξη ενός συστήματος βαθμολογίας πράσινης για τα κτίρια, το οποίο ξέρετε βοηθάει για την ανάπτυξη των βιώσιμων κτιριών, όπου οι αρχές και η ΟΤΑ μπορούν μέσω της ενίσχυσης των κανόνων να αυξήσουν ακριβώς αυτή την ενεργειακή απόδοση των κτιριών. Αυτοί είναι δύο λοιπόν κύριοι τομείς, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλους, αλλά να σας δώσω σύντομα κάποια παραδείγματα. Η ενέργεια και η ΟΤΑ. Ας πάρουμε το Αμβούργο σαν παράδειγμα, όπου έγινε ένα δημοψήφισμα για, για το δίκτυο ενέργειας, το οποίο επαναδημοτικοποιήθηκε το οποίο αποδεικνύει ακριβώς πόσο μπορεί να συμμετάσχουν οι ΟΤΑ στα δίκτυα και στη διανομή ενέργειας, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν είχαν έλεγχο Η Διαχείριση απορριμμάτων αναφέρθηκε και αυτό και αυτό ήταν επίση πολύ σημαντικό. Ένα παράδειγμα τη Φιλανδία εδώ, όπου δημιουργείται ενέργεια, μειώνονται οι εκπομπές ταυτόχρονα, οι εκπομπές που προέρχονται από το χιτά μέσω χρήσης αερίου. Βεβαίως μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική και πιο βιώσιμη η μείωση των εκπομπών. Αν δούμε εδώ ένα παράδειγμα στη Στοκχόλμη, όπου έχουμε μια πρώην βιομηχανική περιοχή, η οποία αναπτύχθηκε με πολύ σημαντική μείωση εκπομπών θερμοκηπίου με πολύ σημαντική μείωση ανακεφαλή σε αυτό το κομμάτι τη ε, πόλη και βεβαίω συνολικά η μείωση ήταν πολύ ε, σοβαρή αν συνδυάσουμε και του τρει τομεί. Βέβαια και η προσαρμογή είναι πολύ σημαντικό πεδίο δουλειά στι τοπικέ αρχέ, στου στόχου τη βιωσιμη ανάπτυξη, ένα μόνο μιλά για το 2020, 2030, 2020 και θεωρούν τι πόλει να προσαρμόσουν τι πολιτικέ του και να προσαρμοστούν στην αντοχή κάτι το οποίο δείχνει δηλαδή τον επίγοντα χαρακτήρα, όπως εδώ στις κάτω χώρες, ε, για την αντιμετώπιση ακριβώς και τη δημιουργία χώρου και περιθωρίου για τους ποταμούς για υπερχείληση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά λοιπόν και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε μια περίπτωση εδώ στον Ειρηνικό, στα νησιά Σολομών, Σολομόντα, όπου εφαρμόζουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής και αυτό να αναπτύσσουν ταυτόχρονα Εθνικέ και τοπικές αρχές ακριβώς για να προστατεύσουν τις ευάλωτε περιοχές, τους πληθυσμού και τους διαφόρους ε, τομεί τη οικονομίας. Συμπεράσματα. Το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε ασφάλεια είναι ότι πραγματικά αυτά τα τρία θεματολόγια εξαρτώνται και αλληλονισχύονται. Ότι είναι καλό για το κλίμα, είναι καλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και καλό για το αστικό θεματολόγιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε σχέση με τα συμπεράσματα των προηγουμένων ετών, δηλαδή καλό για τις πόλεις και για το περιβάλλον και για την κοινωνική διάσταση και για την οικονομική διάσταση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω έβριμα το οποίο μπορούμε να προβάλλουμε και το οποίο μπορεί να βοηθήσει τα άλλα δύο θεματολόγια. Το δεύτερο είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί, θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια ριζόντια ενσωμάτωση. Δηλαδή θα πρέπει τα ξεπεράσουμε τα τοπικά όρια, γιατί πολλέ από αυτέ τι δράσει τι τοπικέ δεν σταματάνε στα τοπικά όρια, όπω η προσαρμογή των οικοσυστημάτων, βιώσιμε μεταφορέ, ε, διαχείριση απορριμμάτων. Όλα αυτά είναι ε, διαδημοτικοί τομεί, διαδημοτικέ προσεγγίσει, όχι δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένε πόλει. Επόμενο συμπέρασμα είναι ότι μία κάθετη ενσωμάτωση αποτελεί ένα προαπαιτούμενο για σημαντική δράση για την καταπολέμηση τη χρηματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ε, κάτι το διτό, δηλαδή αφενό έχουμε κάτι το οποίο ε, πηγαίνει από το εθνικό στο τοπικό, ώστε να ενισχύσουμε ακριβώ του ΣΟΤΑ για να δημιουργήσουν πλαίσια ώστε να προσεγγίσουν του πολίτε, αλλά επίση από το τοπικό στο εθνικό, επειδή η τοπική πρόσφαση θα πρέπει να είναι ε, μετρήσιμη και επαληθεύσιμη. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για μια πραγματική κλιματική δράση και αποτελεσματική. Τέλος θεωρούμε ότι το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο ξεκίνησε φέτος, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να ενθαρρύνουμε πιο φιλόδοξες κλιματικές δράσεις. Όπως ξέρετε, αποτελεί ένα συγκέρασμα ευρωπαϊκών και άλλων παγκοσμίων πρωτοβουλειών, δημάρχων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7.000 πολίτες που εκπροσωπούν 650 εκατομμύρια κατοίκους και που έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν προγράμματα άμβλησης της κλιματικής αλλαγής και να σχεδιάζουν για ευρύτερη και μεγαλύτερη υπερβολική δράση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα με την ε, παρουσίαση από πλευρά τη κυρία Αλεξάνδρα και Ελπίζω να φέρα σωστά το όνομά σα σε ό,τι αφορά την ε, προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Η κυρία Κασμίρσα είναι project manager σε ό,τι αφορά την ε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σε ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνετε να προφέρετε σωστά το όνομά μου, γιατί είναι πάντοτε δύσκολο να το προφέρει κανένας. Σε αυτή λοιπόν την παρουσίαση που θα σας κάνω θα αναφερθώ στον αντίκτυπο της κλιματικής ε, μεταβολής που βλέπουμε στις πόλεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι ακριβώς σημαίνει για αυτές. Στη συνέχεια θα αναφερθώ εν συντομία στο πού βρισκόμαστε ως προς τον βαθμό δηλαδή προσαρμογής των ευρωπαϊκών πόλεων στην κλιματική αλλαγή και μετά θα πω δύο λόγια σε ό,τι αφορά ε, τις πληροφορίε και τις εκθέσεις από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Δημονισμού Περιβάλλοντος και θα κλείσω την παρουσίαση με κάποιες προκλήσεις σε ό,τι αφορά αυτή την προσαρμογή των πόλεων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ διαφοροποιημένες επιπτώσεις ανάλογα με την κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, στο Νότο και ε, γενικότερα ε, στην υπηρετική Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, δασικών πυρκαγιών, ξηρασίων, όπως είδαμε για παράδειγμα και πολύ πρόσφατα τώρα στην Πορτογαλία τις πυρκαγιές. Αντιθέτω, τώρα στην βόρειο-δυτική Ευρώπη αναμένουμε περισσότερε πλημμύρε και ξαφνικέ πλημμύρε, δηλαδή από απότομε και ισχυρότατε βροχοπτώσει, αλλά και από ποταμού πλημμύρε. Άρα λοιπόν τι μας δείχνει αυτός ο χάρτης ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχει ιδιαίτερα τοπικό χαρακτήρα και αυτή η τοπική διάσταση θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη για να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων κλιματικών συνθήκων. Όμως ταυτόχρονα μας δείχνει αυτός ο χάρτης ότι υπάρχουν μεγάλες περιοχές οι οποίες ε, ε, θα αρκεθούν να αντιμετωπίσουν παρόμοια κλιματικά φαινόμενα οπότε αυτό δείχνει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να βρουν τρόπους να συνεργαστούν μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Τώρα, γιατί εστιάζουμε ειδικότερα στι ε, πόλει. Γιατί στι πόλει έχουμε ε, υψηλέ φυσικά συγκεντρώσει πληθυσμού, αλλά και ε, οικονομικών και πολιτισμικών αγαθών, τα οποία βέβαια είναι πολύ πιο ευάλωτα και σε ζημίε. Αλλά από εκεί και μετά η ίδια η σύσταση των πόλεων επιτείνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επειδή δηλαδή είναι σχετικά απομονωμένες αν θέλετε περιοχές σημαίνει ότι θερμοκρασίες τη πόλης είναι πιο αυξημένες και σημαίνει επίσης ότι ε, το ε, νερό των πλημμύρων συγκεντρώνεται εκεί και δεν έχει τη δυνατότητα να ε, διαφύγει, να απορρέψει δηλαδή άλλο. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά τόσο εκτεταμένες, εκτεταμένα τέτοια καιρικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, ο καύσωνας στον Αύγουστο του 2003 προκάλεσε 70.000 θανάτους σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ βέβαια η πλειοψηφία αυτών των Ατόμου που έχασαν τη ζωή του ε, γέμεναν σε πόλει. Από εκεί και μετά είχαμε τι ξαφνικέ πλημμύρε ε, στη Γένοβα του 2014, όπου ε, μέσα σε δύο ώρες έπεσαν 15 εκατοστά βροχή με αποτέλεσμα να ε, δημιουργηθούν ε, ζημίες στις τάξεις των 100 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ λοιπόν έχουμε να, να κάνουμε με τέτοιου είδους φαινόμενα ακραία τα οποία αναμένουμε πως θα γίνουν ακόμα πιο συχνά και ακόμα πιο ακραία στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι πόλεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και μάλιστα αυτό είναι επίγον όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Σημαίνει Κατά συνέπεια ότι οι πολίτες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις αναμενόμενες αυτές τις αλλαγές. Και πώς θα γίνει η προσαρμογή από την πλευρά των πολιτών στην έκθεση της, ε, ως έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ε, αναφέρεται σε τρία είδη προσαρμογής. Ε, καταρχήν στην γκρίζα υποδομή, δηλαδή της πιο αρχιτεκτονικού χαρακτήρα παραδοσιακές λύσεις. Μετά πράσινη υποδομή, δηλαδή χώρους πρασίνου αλλά και χώρους συγκέντρωσης νερού που μπορούν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν τις πιέσεις που ασκούνται στις πόλεις ειδικότερα από τις επλημμύρες και μετά μαλακού τύπου όπως λέγονται soft προσεγγίσεις όπως για παράδειγμα ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των επιπτώσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα το πού βρισκόμαστε ω προ την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη. Η εν λόγω στρατηγική για την ε, ε, προσαρμογή υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το 2013 και βασίζεται σε τρει στόχου. Προώθηση δράσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, προώθηση ε, καλύτερη, πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων. Και τρίτον, προώθηση τη ε, προσαρμογή σε κύριους ευάλωτους ε, τομείς. Ε, σε ό,τι αφορά τα, τις δράσεις από την πλευρά των κρατών μελών, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή 23 από τα 28 κράτη-μέλη έχουν ήδη οθετήσει τις εθνικές τους στρατηγικές για την προσαρμογή και από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά το επίπεδο των πόλεων, το, όπως ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής, το Σύμφωνο των Δημάρχων ξεκίνησε μια πρωτοβουλία το 2014 με την ονομασία Δήμαρχη, η Δήμη ε, προσαρμόζονται. Και από το 2017 και μετά έχει λάβει πιο παγκόσμιο χαρακτήρα αυτή η πρωτοβουλία. Ε, όπως αναφέρθηκε ήδη, το 20% του συνόλου των, της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά επίσης υπάρχουν και ε, μεγάλες προσπάθειες που γίνονται, για παράδειγμα στο πλαίσιο του Horizon 2020, ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας. Αλλά και μέσω του LIFE αντίστοιχε επενδύσει γίνονται στο τομέα τη έρευνα. Από εκεί και μετά και στο πλαίσιο του δεύτερου στόχου, δηλαδή την προώθηση τη καλύτερη ε, ενημέρωση ε, υψηλότερη ευαισθητοποίηση, εδώ λοιπόν ο οργανισμό. Ε, ε, έχει εκπονήσει μία σειρά από εκθέσεις ε, και παρέχει πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ε, βιωσιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα ευάλωτα σημεία σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής. Μία από τις υπηρεσίες του οργανισμού περιβάλλοντος συντηρεί μία κοινή ιστοσελίδα με τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα ε, μια πλατφόρμα λοιπόν η οποία υποστηρίζει τις ε, στρατηγικές πολιτικές και δράσεις ε, προσαρμογής. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα αστικά ζητήματα, περιλαμβάνει εν λόγω πλατφόρμα συγκεκριμένες case studies, δηλαδή περιπτωσιολογικές μελέτες και παρέχει και βήμα προς βήμα καθοδήγησης για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ως προς το πώς να αναπτύξουν τις στρατηγικές για την προσαρμογή τους. Επίσης περιλαμβάνει και γύρω στα 100 προφίλ πόλεων, ε, των ε, πόλεων δηλαδή ε, που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Επίσης, στην τελευταία μας έκθεση εξετάσαμε την προσαρμογή για το τι έχει επιτευχθεί σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής από το 2012 και μετά. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει πράγματι η ανάληψη δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της πόλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βρισκόμαστε κυρίως στο πλαίσιο του σχεδιασμού ακόμα. Δηλαδή η εφαρμογή των λόγων στατιστικών, ε, στρατηγικών έχει αρχίσει μόνο σε ορισμένες πόλεις. Ε, όπου έχουμε τέτοιου είδους σχέδια προσαρμογής ε, ε, προτιμώνται αυτές οι μαλακού soft προσεγγίσεις, μαλακού τύπου προσεγγίσεις, όχι δηλαδή μέσω θέσπισης κανονισμών και επίσημων πολιτικών. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση σε λύσεις που βασίζονται σε φυσικά, σε, στη φύση, δηλαδή πράσινου τύπου, σε ό,τι αφορά δηλαδή περιοχές συσσόρευσης των νερών και ούτω καθεξής. Εκείνο ε, που είναι δηλαδή σημαντικό είναι να υπάρχει ε, μια πιο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση ό,τι αφορά τις λύσεις προσαρμογής και δεν θα πρέπει να είναι κοντόφθαλμες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των πόλεων προκειμένου να είναι προετοιμασμένες για την κλιματική αλλαγή. Ε, σε αυτούς εδώ τους ε, χάρτες βλέπουμε στα αριστερά τον αριθμό των όλων ε, που, συμμετείχαν ε, το 2015 προς υπέγραψαν το, την πρωτοβουλία City το 148 λοιπόν πόλεις, στα τέλη του 2015 και ακριβώς για να σας δείξω το ποια είναι η πρόοδος που επιτεύχθηκε, τον Ιούνιο του, στις αρχές του Ιουνίου του 2017 πάνω από 700 ε, αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης είχαν προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και 900, 900 ε, οργανισμοί σημαντικά στο, στο, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής ε, ε, Υπήρου. Ε, και από εκεί και μετά στο δεξί χάρτη, δεξιό χάρτη βλέπετε την συμμετοχή των πόλεων ε, σε διάφορες παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Αυτός ο χάρτης μας δείχνει δεδομένα από το 2015, οπότε είναι λίγο παροχημένος, αλλά βλέπουμε εδώ τεράστιες διαφορές σε ό,τι αφορά την γεωγραφική κατανομή της συμμετοχής. Δηλαδή υπάρχουν Συγκεκριμένε πόλεις, σε συγκεκριμένε περιοχές που συμμετέχουν σε τέτοιου είδου διεθνεί ε, πρωτοβουλίε, για παράδειγμα η Βαρκελόνη, το Παρίσι και άλλε. Τώρα, ποια είναι κάποια παραδείγματα προσαρμογών. Ε, βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα από την ε, Κοπεχάγη. Μετά δηλαδή από την εξαφνική πλημμύρα του 2011 δημιουργήθηκε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των ξαφλικών αυτών καταιγίδων και ε, αποφασίστηκε να εφαρμοστούν ε, κατά τη διάρκεια 20 ετών 30 διαφορετικά έργα για την αντιμετώπιση αυτών των ε, ε, ξαφνικών ε, καταιγίδων. Ε, κάποιες από αυτές, κάποια αυτά τα έργα λοιπόν έχουν αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, αλλά πολλά από αυτά στοχεύουν στην αλλαγή του αστικού χώρου και, την, και το περισσότερο πράσινο. Για παράδειγμα βλέπετε αυτή την πλατεία η οποία είναι πιο πράσινη. αποτέλεσμα να δίνει μια δυνατότητα στα νερά να απορροφηθούν αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αξιοποιηθεί από τον πληθυσμό και για κοινωνικούς σκοπούς. Προφανώς η προσαρμογή ε, μιας πόλης σε τέτοιο μαζικό επίπεδο είναι κάτι το πολύ δύσκολο ε, και απαιτεί ε, και τα κατάλληλα τα απαραίτητα κονδύλια. Για παράδειγμα για τα 20 έτη Κοπεχάγη έχει προσβλέψει 1,9 δις ευρώ. Οπότε ένα από του στόχου τη εκθεσή μα είναι ακριβώ το να διερευνήσουμε το πώ μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων. Εδώ έχουμε περιπτωσιολογικέ μελέτε από 11 πόλει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αποτελούν ε, βέβαια ε, περισσότερο ένα είδο έμπνευση για το τι μπορούν να κάνουν οι πόλει και όχι μια γενική επισκόπηση του τι συμβαίνει. Πάντω το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να είναι δύσκολο για τι πόλει να βρουν την κατάλληλη χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση των σχετικών τράσεων, αλλά ακόμα και όταν μπορούν να βρουν την κατάλληλη χρηματοδότηση, από, για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι πόλεις δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να προβούν στην υποβολή τη αίτηση. δηλαδή να αξιώσουν ακριβώ σχετική χρηματοδότηση. Ένα ακόμα συμπέρασμα ήταν ότι η συμπερίληψη της πτυχής ακριβώς της κλιματικής προσαρμογής στις απαιτήσεις για παράδειγμα για νέες επενδύσεις θα εξοικονομήσει πόρους αλλά βέβαια αυτό θα γίνει και σε μόνο ε, μακροπρόθεσμα από εκεί και μετά θα πρέπει ε, ε, να καταδειχθεί καλύτερα ε, ε, ο μεγάλος αριθμός πλεονεκτημάτων που μπορεί να επιτευχθεί μέσω ε, των λύσεων προσαρμογής, όπως σας είπαμε για παράδειγμα με το περισσότερο πράσινο στις πόλεις. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε συνολικά ότι οι κύριες προκλήσεις είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι είναι πρωτεργάτες της πόλης, δηλαδή που κάνουν πολλά, και τις πόλεις εκείνες που ακόμα δεν συμβαίνουν πολλά. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ανταλλαγής γνώσεων, αλλά και μέσω εφαρμογής έργων προγραμμάτων των Ιντερεκ, για τα οποία θα ενημερωθούμε σε λίγο, αλλά και μέσω τη κατάλληλη χρηματοδότηση. Δηλαδή και περισσότερε πηγέ χρηματοδότηση, αλλά και τρόπου για πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση για τι πόλει. Από εκεί και μετά, κάτι που ακόμα θα πρέπει να κάνουμε είναι να ε, υιοθετήσουμε μια μετασχηματιστική ε, προσέγγιση ό,τι αφορά την προσέγγιση. Δηλαδή να αλλάξουν ε, οι πόλεις, ε, τα συστήματα διακυβέρνησή του, να αλλάξουν του αστικού χώρου την αστική ρημοτομία, προκειμένου ακριβώ να προετοιμαστούν για τα μελλοντικά καιρικά φαινόμενα. Επίση, θα χρειαστεί καλύτερη ανάπτυξη και συντήρηση του υποστηρικτικού πλαισίου διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή ευρωπαϊκό, ενωσιακό, εθνικό και τοπικό και επίση εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο ε, με ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, είναι και κοινωνικό πρόβλημα, γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή των ε, πολιτών που διαμένουν στι ε, πόλει. Με αποτέλεσμα δηλαδή να θέλουμε να του προστατεύσουμε και από τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή. Η τελευταία πρόκληση είναι ότι οι πόλεις χρειάζονται πολύ καθοδήγηση ω προ το πώ θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα και ακριβώς το πόρταλ που σας παρουσίασα παρέχει τις σχετικές ε, πληροφορίες για την καθοδήγηση. Ε, παρότι αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, το να κατευθυνθούν προς τα εγγύη οι πόλεις και να λάβουν την κατάλληλη χρηματοδότηση παραμένει ακόμα ως ε, πρόκληση στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με την παρουσίαση της κυρίας Κριστιαν Μπρέσνιγκ που είναι επικεφαλής της διαχειριστικής αρχής της πόλης της Βιέννης όσον αφορά το Ιντερεκ για την Κεντρική Ευρώπη. Θα μας εξηγήσει πώς η διαμεθοριακή συνεργασία βοηθάει τις πόλεις να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Από την εμπειρία τουλάχιστον του Ιντερεκ στην Κεντρική Ευρώπη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να σας παρουσιάσω σήμερα τι συμβαίνει στις πόλεις της κεντρικής Ευρώπης όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια από διαμεθοριακά προγράμματα προκειμένου να βρεθούν κατάλληλες λύσεις. Η σημερινή μου παρουσίαση χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα σας παρουσιάσει τα προγράμματα διαμεθοριακής συνεργασίας και πώς αυτά ενσωματώνονται στα διορθωτικά κονδύλια. Και μετά θα σας δώσω τέσσερα παραδείγματα από 27 προγράμματα που έχουμε για το πώς οι πόλεις αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή. Μα ζητήθηκε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε μεσαίες και μικρές πόλεις. Οπότε τέτοια παραδείγματα έχω επιλέξει κι εγώ. Άκουσα και τις παρουσιάσεις βέβαια των προηγούμενων ομιλητών και νομίζω ότι η δικιά μου παρουσίαση όντω συνδέεται πολύ καλά με συμπεράσματα και πληροφορίες που μας έδωσαν οι προλαλήσαντες. Ίσως να γνωρίζετε αυτό το πίνακα, είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας παρουσιάζει λιγάκι ποιο είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, που είναι σχεδόν 3% του προϋπολογισμού της ε, συνοχής. Χρήματα τα οποία μοιράζονται 15 προγράμματα. Αυτά είναι τα 15 προγράμματα εδώ. Η Κεντρική Ευρώπη, βλέπετε εδώ, το δικό μου το πρόγραμμα είναι στη μέση, είναι αυτό το κόκκινο, αυτό διαχειρίζομαι. Τα διαμεθοριακά προγράμματα μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές σχέσεις για να αποτελέσουν στοιχείο μοχλό σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Τα προγράμματα, κάθε πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τέσσερις θεματικούς στόχους. Κάτι που ανέφερε και ο κύριος Νέσπιτ νωρίτερα. Η Κεντρική Ευρώπη λοιπόν αποφάσισε να επιλέξει ως μια προτεραιότητα την, το στόχο 4 που είναι χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και υπάρχουν και άλλες 6 που εδώ πλησιώνονται με κόκκινο που έχουν επιλέξει τον ίδιο στόχο. Αυτό για να σας δείξω ότι στην δικιά μας περιοχή ο στόχος αυτός αποτέλεσε μεγάλη προτεραιότητα. Τώρα τι γίνεται με τα διαμεθοριακά προγράμματα γενικά, μια που δεν έχουμε τα περισσότερα χρήματα εμείς όπως βλέπετε. Οπότε δημιουργούμε στρατηγικές, προγράμματα δράσης, πιλωτικά προγράμματα. Προσπαθούμε εμείς να αρχίσουμε με κάποιες ιδέες οι οποίες θα επεκταθούν περισσότερο στη συνέχεια. Και δίνουμε και πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε πολλά Επίπεδο διακυβέρνησης. Πολλαπλά επίπεδα. Τώρα, τι γίνεται εδώ στην Κεντρική Ευρώπη. Εδώ έχετε τα νούμερα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Τα έχετε και στο τραπέζι. Έχουμε εννέα ε, συμμετοχές σε κράτη-μέλη, 150 εκατομμύρια ε, πολίτες, καλύπτουμε 250 εκατομμύρια για 7 χρόνια. Και αυτό που είναι Πιο σημαντικό ακόμα και από αυτά τα στοιχεία είναι ότι στους δύο διαγωνισμούς που ήδη έγιναν απορροφήσαμε 70% ήδη των κονδυλίων και από τους 900 εταίρους που χρηματοδοτούμε 200 είναι πόλεις. Άρα είναι πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε την πρώτη περίοδο 2007-2013. Αυτό όμως που επίσης πρέπει να πούμε τώρα είναι ότι στις δύο αυτές προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος, πάνω 50% πήγανε σε προγράμματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Χάρη στους κώδικες αυτούς παρέμβασης, το εκτιμάμε αυτό, και μπορούμε πιο εύκολα πια να πούμε πόσο συνεισφέρουν τα προγράμματα αυτά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για αυτήν την διαφάνεια, αλλά εδώ σας εξηγούμε ότι δεν υπάρχει μόνο η οικονομία χαμηλού άνθρακα ως προτεραιότητα, υπόθηκε αυτό και νωρίτερα, έχουμε το περιβάλλον, ο θεματικός στόχος 6 δηλαδή είναι πολύ σημαντικός και τον χρηματοδοτούμε πολύ στα προγράμματά μας. Κάποια άλλα τώρα σημαντικά στοιχεία, γιατί έχουμε τόσο πολλές πόλεις που ζητούν χρηματοδότηση. Η Κεντρική Ευρώπη διαθέτει εκατοντάδες μικρούς δήμους, πάρα πολλές πόλεις μεσαίου μεγέθους και αν βάλουμε μέσα και την Κροατία που συμμετέχει αυτή στο πρόγραμμά μας, έχουμε επτά πρωτεύουσε. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια ομάδα στόχο για μας και μας επιτρέπει να συνδυαστούμε και με την Ήπεθρο εφόσον οι πόλεις που εμείς χρηματοδοτούμε συνδέονται με κάποιο τρόπο και με την Ήπεθρο. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η δυνατότητα προσαρμογής των πόλεων στην κεντρική Ευρώπη. Ο χάρτης αυτός δείχνει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των περιοχών μας Βλέπετε εδώ πώς γίνεται η διάκριση ανάμεσα στις περιοχές εκείνες που βρίσκονται δεξιά από το παλιό σιδηρούν παραπέτασμα που γνωρίζουμε και τι γίνεται στην άλλη μεριά. Λοιπόν, έχετε στο μυαλό σας αυτή την εικόνα, συνδυάστε την και με αυτήν την εικόνα που σας δείχνω τώρα, που δείχνει πόσο ευάλωτες είναι αυτές οι περιοχές που έχουν πολύ μικρή δυνατότητα προσαρμογής για να να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούν να επενδύσουν σε μέτρα ε, προσαρμογής ή μετριασμού των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Όπως είπε επίσης και η κυρία Κασμίρτσακ, στις περιοχές αυτές έχουμε κυρίως πρόβλημα έλαψης ύδατος μερικές φορές ή αντίθετα πλημμυρών. Έχουμε δηλαδή πολλές ακραίες περιπτώσεις να αντιμετωπίσουμε. Η ανταγωνιστικότητα και το ΕΠ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορεί κανείς να προσαρμοστεί ή να είναι λιγότερο ευάλωτος. Οι πόλεις όμως δεν μπορούν να περιμένουν. Είναι δραστήριες στην κεντρική Ευρώπη, δραστηριοποιούνται, γιατί οι δήμαρχοι δεν μπορούν να περιμένουν, ξέρουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Και αυτή εδώ η εικόνα νομίζω ότι δείχνει καλύτερα από οποιοδήποτε κατάλογο που θα μπορούσα να σας παρουσιάσω πώς χρησιμοποιούν οι πόλεις το πρόγραμμά μας, γιατί προβλέπει συνεργασία, χρηματοδότηση, know-how, ανταλλαγές και μεταφορά βέλτιστων πρακτικών. Αυτή είναι μια εικόνα από την περίοδο 2007-2013 και δείχνει πόσο συνδέονται 270 εταίρε 26 προγράμματα που έχουν να κάνουν μόνο με την κλιματική αλλαγή, όχι με μεταφορές, καινοτομία ή άλλα. Πιστεύουμε ότι αν βάλουμε μέσα και άλλα προγράμματα θα είναι ακόμα πιο δυνατή η εικόνα στην οποία θα καταλήγαμε. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η στενή συνεργασία και βλέπετε ότι συμμετέχουν και κάποιες πόλεις και περιοχές εκτός της περιοχής του προγράμματος. Έρχομαι τώρα στα παραδείγματα. Πόλεις και πώς προσαρμόζονται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε ακούσει πολλά για αυτό που ονομάζουμε ε, UHI, Urban Heat Islands, δηλαδή πόλεις και πώς θα αντιμετωπίσουν την ε, αύξηση της θερμοκρασίας πώς θα βελτιωθούν επίσης οι συνθήκες ζωής στις πόλεις αυτές. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει και δικιά μου η πόλη, η Βιέννη και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μπορείτε να διαβάσετε στις πληροφορίες που σας έχω δώσει, πώς συνδέονται οι πόλεις και τι κάνουν, πώς συνεργάζονται και τα είπε και ο σας, τι πρωτοβουλίες μπορεί κανείς να πάρει. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε την οριζόντια συνεργασία. Δηλαδή συνεργάζονται οι πόλεις μεταξύ τους, συμπεριλαμβάνονται και λειτουργικές ε, περιοχές, συνεργάζεται το τοπικό επίπεδο αλλά και το εθνικό επίπεδο σε πολυτομιακές συνεργασίες. Έχουμε περιβαλλοντολόγους, πανεπιστήμια, ε, σχεδιαστές ε, χωροταξίας κλπ. κλπ. Το δεύτερο παράδειγμα δεν έχει να κάνει με την προσαρμογή, έχει να κάνει περισσότερο με το μετριασμό των επιπτώσεων. Και η ομάδα στόχος είναι πολύ μικρή δήμη που δεν διαθέτουν το know-how, αλλά δεν έχουν ούτε και την ικανότητα να εφαρμόσουν προγράμματα ενεργειακού σχεδιασμού ή ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για 34 πόλεις που συνεργάστηκαν στο πρόγραμμα αυτό που το ονομάσαμε Manergy. Και αυτό προκειμένου να εκπονηθούν σχέδια ενεργειακής απόδοσης και να δημιουργηθούν ενεργειακές υπηρεσίες. Εδώ, αυτοί οι δήμοι δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν την γνώση από μόνες τους αν δεν είχαν τη δυνατότητα συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα βλέπετε και ποιος είναι ο προπολογισμός, 1,1 εκατομμύριο για 34 πόλεις. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό είναι ότι στο πρόγραμμα μας εδώ τα καλύτερα αποτελέσματα τα βλέπουμε συνήθως μετά. Δηλαδή δημιουργείται εδώ ένα φαινόμενο μόχλευσης, διότι προσελκύονται επενδύσει, όπως έγινε και σε αυτή την περίπτωση, για την μόνωση των κτηρίων, για φωτοβολταϊκά κλπ. Επιπλέον, οι 21 από αυτούς τους Δήμους συμμετείχαν στη συνέχεια και στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων. Επόμενο παράδειγμα. Πάλι για τον μετριασμό των επιπτώσεων και έχει να κάνει και με την ενεργειακή απόδοση σε δημόσια κτίρια. Εδώ συμμετέχουν πόλεις, δήμοι, συνεργάζονται μεταξύ τους και έφτιαξαν 7 εμβληματικά κτίρια που αποτελούν το παράδειγμα. Και έφτιαξε και καινούρια κτίρια. Δεν μετέτρεψαν μόνο παλιά. Και υπάρχει και ένα πρόγραμμα αξιολόγησης βιωσιμότητας κτίριων, όπου μπορεί κανείς να βρει κριτήρια ώστε να μπορέσει να ελέγξει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων πολύ εύκολα με μια εφαρμογή online. Τώρα ποια είναι η γεωγραφική κατανομή. Είναι από την Ανατολή στη Δύση, από βορρά στο Νότο, για να συμπεριληφθούν ακριβώς και οι περιοχές εκείνες που είδατε πριν στο χάρτη και που θεωρούνται άκρος ευάλωτες και που πιο δύσκολα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Το τελευταίο πρόγραμμα που θέλω να σας παρουσιάσω και θα κλείσω με αυτό, έχει να κάνει πάλι με το μετριασμό των επιπτώσεων. Δεν έχει να κάνει με νέα κτίρια, έχει να κάνει με ήδη υπάρχοντα κτίρια. Και εδώ πώς θα διαχειριστούμε με πιο έξυπνο τρόπο την ενέργεια. Εδώ είχαμε πάρα πολλές αιτήσει όταν προκυρήσαμε ε, τα προγράμματα αυτά. Προς το παρόν θα βρείτε και υλικό εδώ στην αίθουσα για να έχετε περισσότερες πληροφορίες αν θέλετε, αλλά μπορείτε να πάτε και στην ιστοσελίδα μας. Πάντως, για αυτούς ε, που είσαστε από περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θέλω να σας πω να ξέρετε ότι θα υπάρχει νέα ε, προκήρυξη για πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος 21 και 22 Σεπτεμβρίου του 2017 για νέο πρόγραμμα. Και ευχαρίστως αν έχετε χρόνο να σας δώσω τη διάσκεψη αυτή, στην οποία θα γίνει αυτή η προκήρυξη, που θα γίνει στο Βερολίνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρουσιάσεις σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους της Κομισιόν να σχολιάσουν και ενδεχομένω να υποβάλουν προτάσεις. Καταρχάς κυρία Γεργάνα Μιλαντίνοβα, υπεύθυνη του Κέντρου Εφιούς και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει το λόγο, κύριε Μιλαντίνοβα. Πρώτα ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για διοργάνωση αυτού του καλού εργαστηρίου. Δύσκολο το έργο μου γιατί είχαμε τόσο καλές εισήγησει. και είναι ενδιαφέρον να δούμε που αυτός ο νέας τομέας, νέος τομέας του κλίματος, νέος μέχρι πρόσφατα, έχει γίνει το επίκεντρο των πολιτικών συνοχής. σε σχέση με τους στόχους. Και πραγματικά ό,τι αφορά το χαμηλό άνθρακα είναι γύρω στο 50%, τουλάχιστον 50%. Και βεβαίω βλέπουμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες προωθούνται μέσω της νομοθεσίας για το, την ενέργεια, μέσω αντιμετώπιση κινδύνου κλπ. κλπ. Έχουμε βεβαίω και το Ίντερεκ και διάφορα άλλα εργαλεία που μας βοηθούν. Έχουμε πετύχει πολλά σε σχέση με την περίοδο 14-20 όσον αφορά την πρόθεση αυτού του ζητήματος. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και απαιτήσει διατομιακές, δηλαδή που αφορούν τις υποδομές, τις μεταφορές, την προσαρμογή την κλιματική και τα αντίστοιχα μέτρα. Οπότε έχουν θετικό αποτέλεσμα αυτές οι δράσεις και συνεχίζονται. Ένα νέο στοιχείο εδώ τώρα είναι οι πόλεις. Μέχρι τώρα είχαν το 5% των κονδυλίων. Πήγε στο 8%. 15 δις θα πάνε στις πόλεις συνολικά. Το 40% αυτό των 15 δις θα πάνε για δράσεις χαμηλού άνθρακα. Και αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα που έχει επιλεχθεί για τις πόλεις. Μετά οι υπόλοιπε ε, προτεραιότητες αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και αυτό είναι ενδεικτικό της αλλαγής στη φύση της πολιτικής συνοχής ή των πολιτικών συνοχής και τη στόχευση στην κλιματική αλλαγή και στην καταπολέμησή της και προστασία του περιβάλλοντος. Θα ήθελα επίσης να τονίσω και το θέμα της εξειδίκευσης και τη έρευνας που γίνεται εκεί από την βιομηχανία ώστε να ρωτήσουν κατάλληλε προτεραιότητε για τις περιφέρειες στα πλαίσια των πολιτικών συνοχής και της προτεραιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το κλίμα. Και το οποίο θα πρέπει για να συνεχίσει να έχει σημασία στο μέλλον να συνοδεύεται από καινοτομία. Γι' αυτό είναι απαραίτητο για να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε να κινητοποιήσουμε την βιομηχανία της έρευνας, αλλά για να έχουμε βέβαια και τα κονδύλια ώστε να επικαιροποιήσουμε αυτούς τους στόχους με τους υπόλοιπους. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε πολλά για τα επιτεύγματα, να μιλήσουμε πολύ για τα επιτεύγματα και υπάρχουν και οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν αναφέρθηκαν οι πόροι, ας πούμε, οι μεθοδολογίες που χρειάζονται και πρέπει να είναι καλύτερες. Αυτό από μόνο το αποτελεί πρόκληση. Είναι ένα τιτάνιο έργο, αλλά βέβαια το ανέφεραν και οι προαλήσαντες, να αναφέρω εγώ και το αστικό θεματολόγιο. Εκτός βέβαια από την ε, στόχευση των κονδυλίων μιλάμε και για άλλες πρωτοβουλίες, δηλαδή την αστική ας πούμε, ατζέντα, το αστικό θεματολόγιο για την Ευρώπη, τους εταίρους που έχουμε εδώ, την κλιματική προσαρμογή, την εταιρική σχέση για τη μετάβαση των μέσων ενέργειας. Να αναφέρω επίσης ότι θα υπάρξει κι άλλος ένας διαγωνισμός, άλλη μια προκήρυξη για την αστική καινοτομία. Υπάρχουν λοιπόν πολλές εξελίξεις και θα ήθελα να τελειώσουμε δύο σημεία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εστιάσουμε στην καινοτομία στις πόλεις αλλά βεβαίω και στα οικονομικά εργαλεία. Στην καλύτερη χρήση τους δηλαδή, ώστε να προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση. Είναι προφανές βέβαια, αλλά ακούγοντας όλα αυτά τα καλά παραδείγματα, νομίζω θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην επικοινωνία. Ξέρω ότι Προσπαθούμε να το κάνουμε και ξέρω ότι είναι σημαντικό να ξέρουν, να γνωρίζουν οι πολίτες τι κάνει η Ευρώπη με τα λεφτά τους. Και θα πρέπει νομίζω να το τονίσουμε ακόμα περισσότερο αυτό. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, λέει Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε με τον Γενικό Διευθυντή από τη Μονάδα Προσαρμογής στη Γενική Διευθύνση για την Κλιματική Δράση, ο κύριος Κλάδος Κόντροπ. Παρακαλώ. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τους συζητητέ για τι εισηγήσεις του Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Σε μία από αυτές ακούσαμε την στρατηγική 2020 και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τους στόχους που αφορούν το μετριασμό των επιπτώσεων. Οι προσπάθειες λοιπόν για το μετριασμό σε αυτό το πλαίσιο εγγράφονται δηλαδή στην προτεραιότητα που ήταν στη στρατηγική 2020. Τώρα έχουμε βέβαια και την επόμενη φάση, 2030, και τη συμφωνία του Παρισιού και την πολιτική συμφωνία για τον μετριασμό. Για την προσαρμογή λοιπόν το οποίο έχει αλλάξει. Αν εξετάσουμε αυτά τα τελικά συμπεράσματα για την περίοδο 14-20, θα δούμε ότι μπορούσαμε να προωθήσουμε τις δράσεις αυτές ε, για το μετριασμό στις, ε, στα κονδύλια που αφορούν και το Ταμείο Συνοχή και το Πεφριακό Ταμείο. Αυτό μας δίνει μια σωστή βάση, μια καλή βάση για περαιτέρω δράσεις. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις, να τις καθοδηγούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά. Βεβαίω, οι πόλει υπόσχονται πολλά εδώ, γιατί είναι πολύ κοντά στον τόπο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και αφορούν ακριβώς τις δράσεις μετριασμού και προσαρμογής. Βλέπουμε εδώ ότι δεν έχουμε να μόνο με πόλεις αλλά και με κομμοπόλεις και παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την μετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Να τελειώσω κι εγώ με δύο λόγια για την στρατηγική προσαρμογής που υιοθετήθηκε το 2013. Βρίσκεται υπό αξιολόγηση τώρα και θα έχουμε μια δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσει στα τέλη του Οκτώβρη, τρίμηνη, τριμηνιαία μάλλον, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, θα είναι δημόσια διαβούλευση και θα έχουμε τα αποτελέσματά τη στα τέλη του έτου στι αρχέ του επόμενου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρο. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Αν έχετε ερωτήσει, προτάσει, σχόλια, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Ροντρίγκες. Ε, δεν έχω να θέσω ένα ερώτημα, απλά ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, που πήραν ε, το λόγο. Εγώ βέβαια είμαι Πορτογαλίδα, οπότε πραγματικά είναι μια ιδιαίτερα ατυχή συγκυρία για μένα σήμερα το να μιλάω για την κλιματική αλλαγή. Είναι... Ε, βέβαια είναι πάρα πολύ ατυχές αυτό και για τους, τον πληθυσμό της χώρας μου. Σε ό,τι αφορά ε, το ζήτημα της ε, ε, πολιτικής βούλησης θα ήθελα να αναφερθώ ότι πολύ συχνά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά και τα ζητήματα της κλιματικής μεταβολής υπάρχει ακριβώς λυπής πολιτική βούληση προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες θα μας είχαν οδηγήσει στο να αποφύγουμε την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Αναφερθήκαμε για παράδειγμα εδώ, ακούσαμε για παράδειγμα ε, ε, κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τις εξόχως ε, απόκεντρες περιοχές. Ε, για παράδειγμα στη δηλαδή στη ε, ε, είδαμε ότι υπάρχουν, υπάρχουν μεγάλα τροτά, αν θέλετε, σημεία τόσο σε ό,τι αφορά ε, όσο και σε ό,τι αφορά πλημμύρες. Οπότε πραγματικά εδώ βλέπουμε πόσο μεγάλε είναι οι προκλήσεις και θα θέλαμε να ακούσουμε από το Ραφάλ, για παράδειγμα, από τον Εθνή, από την Αλεξάνδρα, κατά πόσο, στον λόγο σύμφωνο στο οποίο αναφέρθηκαν, προβλέπεται ε, κάποιο τρόπο για να εφαρμοστεί τελικά η νομοθεσία. νομοθεσία η οποία θα έπρεπε να ε, εφαρμόζεται ε, προκειμένου να προστατευτούν οι πολίτε. Για παράδειγμα, συχνά. για παράδειγμα, δεν τηρείται μια νομοθεσία η οποία υφίσταται στην Πορτογαλία και είναι δεσμευτική σε ό,τι αφορά τον, την αποψήλωση των συγκεκριμένων εκτάσεων. Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη σε ό,τι αφορά τις πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται αλλά και την καλύτερη ευαισθητοποίηση του ε, κοινού και εδώ ε, νομίζω πως θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερο ρόλο οι δήμοι και οι κοινότητες ε, προκειμένου ακριβώς να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επίσης θα ήθελα να ακούσω εάν υπάρχει κάποια δράση η οποία έχει αναλυφθεί ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των εξόχων, εξόχων από ό,τι των περιοχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας ε, για τις παρουσιάσεις που έκανα σήμερα εδώ. Ε, όπως ε, είπε και η ε, προηγούμενη ομιλήτρια, πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ε, ζήτημα για τη δική μα ε, ομάδα και εμεί από την πλευρά των Πρασίνων θεωρούσαμε πω ήταν πολύ σημαντικό να γίνει η σημερινή συζήτηση. Επειδή γνωρίζω ότι έχουμε πίεση χρόνου, θα είμαι πολύ σύντομη. Είναι κοινό μα στόχο να βελτιώσουμε τη συνεισφορά τη πολιτική συνοχή στην επίτευξη των κοινών στόχων για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Η μελέτη του κυρίου Νίσπετ, την οποία μας παρουσίασε σήμερα ε, ε, αποτελεί ένα, ε, μία ακόμα ένδειξη ότι τελικά το 20% των, των, των, της δέσμευσης του προπολογισμού για την κλιματική αλλαγή δεν θα επιτευχθεί τελικά παρά τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί. Και επίσης ένα ακόμα ζήτημα το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι δεν υπάρχει μια σαφής και συνεκτική διαδικασία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ε, παρακολούθηση. Ε, ε, και γνωρίζετε πως εμείς έχουμε από την πλευρά των Πρασίνων πολύ συγκεκριμένες για τις συγκεκριμένες ε, πολιτικές, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά δεσμευτικούς, ε, δεσμευτικά ποσοστά, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ή για παράδειγμα σύνδεση μεταξύ των ε, εθνικών σχετικών προγραμμάτων δράσης και των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων. Οπότε ένα σχετικά, αν θέλετε, απλό ερώτημα από την πλευρά μου είναι το εξής θεωρείτε πως η απλούστερη λύση για την ενίσχυση του mainstreaming ε, των δράσεων για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή την ένταξή του ε, στις βασικές πολιτικές, είναι να προβλεφθούν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις και στόχοι. Και αν ναι, αν πιστεύετε πως αυτή είναι η λύση, η απλούστερη λύση. Ε, ε, πού θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει, στο εθνικό επίπεδο ή στο επίπεδο της εφαρμογή των προγραμμάτων. Και από εκεί και μετά θεωρείται πως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδος μαύρης λίστας σε ό,τι αφορά τις δαπάνες οι οποίες έχουν ανητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Και ε, τέλος, επειδή εγώ κατάγομαι από τη Βιέννη, όπου εδώ βέβαια το αστικό θεματολόγιο είναι πολύ σημαντικό, και αναφέρθηκε εδώ, είναι πολύ σημαντικό και η δική μας Επιτροπή, θα ήθελα να ακούσω κάποιες προτάσεις από τη δική σας πλευρά. Πώς μπορούμε δηλαδή να ενισχύσουμε περισσότερο το αστικά θεματολόγιο προκειμένου να ε, γεφυρώσουμε το χάσμα στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή μεταξύ αυτών των πόλεων που κάνουν πάρα πολλά και έχουν προχωρήσει πολλά, μεταξύ αυτών και η Βιέννη, και των πόλεων εκείνων οι οποίες ακόμα δεν έχουν αναλάβει εκτεταμένες δράσεις σε ό,τι αφορά την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Τεμάτο. ευχαριστώ για τη χρήση της γης. μην φαινόμαστε διπολικοί στους πολίτες, γιατί μιλάμε αφενός για μετριασμό όσον αφορά το, τις επιπτώσεις στα εδάφια και αφετέρου η Κομισιόν στηρίζει πολιτικές οι οποίες αφαιρούν γη από την γεωργία, ιδιαίτερα μέσω πρώτης καυσίμων. Ορυκτών. Οπότε εδώ ποια είναι η πιο αποτελεσματική πολιτική στο τομέα αυτό. Μετά αναρωτιέμαι τι θα γίνει στο μέλλον το ΕΖΕΦ και το ΕΦΣΥ. Γιατί ξέρουμε το ΕΦΣΥ μέχρι τώρα χρηματοδοτεί και στηρίζει τα ορυκτά καύσιμα. Τι θα γίνει με το 20% του ΕΣΥΦ, θα αλλάξει και κλείνουμε ένα σημαντικό ερώτημα προς την Κομισιόν. Ποια είναι η απόψη της για την σύσταση ενός ταμείου όπως στη ΣΥΠΑ από τη βιομηχανία σε σχέση με τις αλλαγές στο, κλίμα, στο περιβάλλον και το κλίμα. Και τι γίνεται ακριβώς με ένα γεωρός που αφορά ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, δηλαδή η ανάκτηση εδαφών που έχουν μολυνθεί από τη βιομηχανία και την επαχρησιμοποίησή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κρέα, η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που κατέφθασα κάπως αργοπορημένη στην ε, συνεδρία σε μας. Ε, θα θέσω ένα ερώτημα ε, ε, για αυτό το λόγο το οποίο ενδεχομένω να έχει ήδη απαντηθεί, αλλά επιτρέψτε μου να το θέσω. Πρόσφατα λοιπόν βρεθήκαμε στο πλαίσιο μιας αντιπροσωπείας ε, εδώ της Επιτροπής μας στις Αζόρες. Και εκεί στην επίσκεψή μας μια ομάδα δημαρχών μας είπε ότι δεν έχει νόημα να δεσμεύουμε το 20% του προπολογισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής, αλλά από την άλλη πλευρά στις Αζόρες να προβαίνουμε για παράδειγμα σε μόνωση κάποιων ε, ε, σπιτιών ε, στις Αζόρες, η οποία παντελώς περιττή αφού ποτέ δεν υπάρχουν θερμοκρασίες κάτω από το 0 στις Αζόρες. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο ακριβείς ήταν αυτές οι περιγραφές από την πλευρά των δημάρχων, πάντως εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Πώ αξιολογείται το δικαίωμα ενεργού συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων από την πλευρά των ε, Δήμων στα κράτη-μέλη. Ποια είναι η εμπειρία σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και δεύτερο, πόσο ευέλικτα μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον ε, στόχο δέσμευση του 20% προπολογισμού. Γιατί βέβαια δεν έχουμε να κάνουμε μόνο εδώ με ζητήματα ενεργειακή απόδοση και μόνωση κτηρίων. Υπάρχουν δηλαδή και άλλε δράσει, άλλοι τομεί στου οποίου μπορούμε να κατευθύνουμε αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Η κυρία Βαλίνα τώρα θα πάρει το λόγο, η οποία είναι η συγγήτριά μα σε ό,τι αφορά την ειδική έκθεση για τον ρόλο των ε, Δήμων και Κοινοτήτων των Πόλεων ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ω ε, προ την εφαρμογή των ε, στόχων ε, για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του εμπειρογνώμονε. Ήταν ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε. Νομίζω Έχουμε πει επανειλημμένω ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενό προβλήματο επίγοντος και διεθνού φύση. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε με την δέσμευσή μα για την καταπολέμηση της κλιματική αλλαγή που αρχίζει να μα πιέζει. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε ως ερετή. Το απαιτεί αυτό όλο και περισσότερο η κοινωνία και οι πολίτες Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να διατηρήσουμε τη θέση μας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των ΗΠΑ από τη συμφωνία μετά από προσωπική απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ που δυστυχώς φαίνεται να ακυρώνει οι διεθνείς συμφωνίες και πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε δεκαετίες δουλειά και προσπαθειών υπέρ του πλανήτη. Νομίζω ότι μια υπερδύναμη αρνούμενη αυτές τις δεσμεύσει της που είναι απαραίτητες για την επιβίωση του κόσμου νομίζω ότι δεν μας ε, βοηθάει και πολύ και δείχνει ένα κακό παράδειγμα. Εμείς λοιπόν ως αιρετοί στα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να είμαστε υποχώρητοι αλλά ταυτόχρονα και ευφυείς να αφορά τις αποφάσεις μας. Και αυτό ακριβώς θεωρώ ότι προετοιμάζουμε αυτή την έκθεση που αποβλέπει ακριβώς στο να συνοψίσει και να ανακατατάξει τις κατευθυντήρες γραμμές διεθνώ και στην Ευρώπη που αφορούν την κατάσταση των περιφερειών όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να εντοπίσουμε απτά μέτρα σε επίπεδο διακυβέρνησης και σε επίπεδο πόρων. Γι' αυτό ακριβώ λοιπόν θέλουμε όχι μόνο να έχουμε στη διάθεσή μας την ανυπολόγιστη βοήθεια πυρογνωμών όπως σήμερα, αλλά επίσης να ξεκινήσουμε διαδικασία ευρεία συμμετοχής των πολιτών, γιατί οι πολίτες έχουν να μας πούν πολλά επ' αυτού, για το πώς θέλουν να ζήσουν, πώς θέλουν να οργανώσουν τις πόλεις τους, σε σχέση με τις μεταφορές τους, με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν, με το είδος ενέργειας που καταναλώνουν. Κατά πόσο αυτό είναι μακρόπνο ή όχι. Νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις, αυτές οι αποφάσεις μας επηρεάζουν καθημερινά. Έχουμε την θέρμανση, του πλανήτη, αλλά εδώ θα πρέπει να ακούσουμε την άποψη των πολιτών για να ανακτήσουμε ακριβώς την εμπιστοσύνη τους, η οποία όλο και χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια συμμετοχική διαδικασία, όχι μόνο με διατομιακού εμπειρογνώμες, αλλά από το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να συμβάλλουμε με ιδέες, με εμπειρίες, με αυτές τι προτάσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο για να δώσουμε και κάποια φύση δυνατή στο κείμενο που προετοιμάσουμε με την συμμετοχή των πολιτών αλλά και για να επικυρώσουμε τις αποφάσεις που θα λάβουμε. Αυτά από μένα, τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή και όλες και αναμένουμε τη συμβολή σας για την έκθεση αυτή και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ και εγώ. Ερωτήσεις. Ποιος θα να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας και μερικές φορές τις δύσκολες ερωτήσεις. Θα αρχίσω από τις εύκολες και ίσως αφήσω τις δύσκολες του συναδέρφους εδώ δεξιά μου. Η κυρία Ροντρίγκε πρώτα απ' όλα ρώτησε για το σύμφωνο των δημάρχων και αν μπορεί αυτό να βοηθήσει καλύτερη εφαρμογή των μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Δεν γνωρίζω αρκετά για την φοβερή τραγωδία στην Πορτογαλία αυτές τις μέρες. Το μόνο που μπορώ βέβαια να σας πω ότι συμπάσχω. Πάντως για τις ερωτήσεις σας, το σύμφωνο αυτό των δημάρχων τι κάνει. Επιτρέπει στους πιο ενθουσιώδεις από τις τοπικές αρχές και τις πόλεις να δεσμευτούν ακόμα περισσότερο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω συνεργασίας μεταξύ των, μέσω της ερεσιμότητας εξάντε για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιφερειακό περισσότερο και σε εθνικό επίπεδο. Η συνοχή σίγουρα ε, βοηθάει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αναφέρατε. Για την κυρία Βάνα. Αναφερθήκατε στην έλλειψη συγκεκριμένης δομής και ανείχνευσης κατά κάποιο τρόπο των προβλημάτων ώστε να δούμε πώς θα φτάσουμε στο 20%. Αυτή η δέσμευση έχει να κάνει με τον συνολικό ευρωπαϊκό Προπολογισμό. και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσουμε το ποσό αυτό στα διάφορα μέσα που διαθέτουμε. Πρώτα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Πρέπει να δούμε βέβαια πώς το βλέπει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα θέλουμε δηλαδή από ποιο ταμείο. Τι θα βάλουμε για την κλιματική προσαρμογή και τι για τον μετριασμό των ε, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Και βέβαια πρέπει να δούμε και πώς το διοικητικό κόστος παίζει μέσα σε αυτά τα κονδύλια και τις δαπάνες για να ξέρουμε ακριβώς πόσα χρήματα πάνε στον κάθε στόχο. Για τις επενδύσεις ναι σίγουρα είναι μια καλή ιδέα το να δούμε και σε άλλες περιπτώσεις αν επενδύσεις σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα σταθμό, πόσο αποτελεσματικά εφαρμόστηκαν, υλοποιήθηκαν. Όντως, θα είχε νόημα αν υπάρχει ένα αρνητικό κατάλογος επενδύσεων. για την κυρία Τομάτο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ναι. Από την εμπειρία που έχουμε από το Superfund στις Ηνωμένες Πολιτείες, μηχανισμοί όπως είναι η εμπορία εκπομπών και πώς χρησιμοποιούνται στη συνέχεια τα δικαιώματα αυτά, Εδώ παίζει ρόλο η πολιτική βούληση που δυστυχώς δεν είναι αρκετή για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε με το σύστημα αυτό εμπορίας εκπομπών. Γι' αυτό λέω ότι αν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιηθούν κονδύλια από αυτό το σύστημα εμπορίας εκπομπών πρέπει να δούμε τι χρήματα θα πάνε σε τι πρόγραμμα. Αυτές θα έλεγα ότι ήταν οι εύκολες ερωτήσεις σας. Τις δύσκολες θα τις αφήσω για τους συναδέρφους. Η κυρία Βαλίνα επικεντρώθηκε βέβαια στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το παράδειγμα που έχουν από διάφορε πόλεις και πολιτείες στις ΗΠΑ που είπαν ότι θα συνεχίσουν να φροντίζουν για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών παρά την αποδέσμευση του Πρόεδρου Τραμπ από το COP21, καταλαβαίνετε ότι κάνει τις προσπάθειές μας ακόμα πιο δυνατές και στέρες. Εντάξει, η σημερινή κυβέρνηση με ενδιαφέρεται λιγότερο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη όμως, οι πόλεις και οι πολιτείες στις Ηνωμένε Πολιτείε δεσμεύονται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επόμενος, για να συμπληρώσω τόσο είπε ο συνάδελφος, όντως το σύμφωνο των δημάρχων δεν είναι δεσμευτικό. Συμφωνήθηκε μεταξύ κάποιων που θέλουν να έχουν ηγετική θέση και ο λόγος είναι ότι οι ρυθμίσεις της πόλης είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο. Πρώτα απ' όλα έχουμε διάφορες ρυθμίσεις οι οποίες είναι ξεπερασμένες. Προσθέτουμε ρυθμίσεις χωρίς να φροντίσουμε να εξαφανίσουμε εκείνες τις οποίες αντικαθιστούν. Όταν μιλάμε για αυτήν την ε, κάθετη ένταξη, δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τα επίπεδα διακυβέρνησης, αλλά πρέπει από το πιο χαμηλό επίπεδο της τοπικής ε, δίκησης να πηγαίνουμε στους πολίτες. Τότε θα λειτουργήσει το σύστημα, να το συμπεριλάβουμε και αυτούς σε αυτή την κάθετη ρύθμιση. Μια άλλη ερώτηση είχε να κάνει με το πώς θα γεφυρώσουμε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με αυτούς που βρίσκονται στο τέλος. Έτσι καλλιώς η προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων είναι κάτι από το οποίο εποφελούνται όλοι. Δυστυχώς όταν υπάρχει μια καταστροφή, όταν διαπιστώνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά, τότε ξεκινάει η προσπάθεια για μια αλλαγή. Όπως επίσης και η φωνή των πολιτών, η κινητοποίηση δηλαδή από πλευρά των πολιτών κινητοποιεί και τους τοπικά εκλεγμένους για να αναλάβουν με τη σειρά τους δράση. Ευχαριστώ. Ωραία. Ποιος θα είναι ο επόμενος? Εσείς παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε αυτό που είπαν οι προηγούμενοι και απαντώντας την κυρία Ροντρίκες Δεν είναι σε θελούσια βάση το Σύμφωνο των Δημάρχων. Όμως οι δήμαρχοι δεσμεύονται για αξιολόγηση των ασθενών σημείων βάσει των στρατηγικών προσαρμογή Οπότε αυτή η δέσμευση σημαίνει τουλάχιστον να γνωρίζουμε μια κατάσταση και τι επιπτώσει που έχει αυτή η κατάσταση στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωή και ότι αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα όχημα προς δράση. Τώρα για το κατά πόσο μπορούμε να καλύψουμε το κενό στην ανταλλαγή των γνώσεων μέσω προγραμμάτων και πρωτοβουλειών όπως αδελφοποίησης κατά πόσο πιο προηγμένες ή λιγότερο προηγμένες ή προχωρημένες πόλεις μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες ώστε να έχουν μια επιτυχή στρατηγική για την κυρία Βαλίνα, για το ρόλο της ε, κοινωνίας των πολιτών. Ναι, έχει τεράστια συμβολή στην στρατηγική προσαρμογή και πραγματικά έχει αναγνωριστεί αυτό όσον αφορά το ρόλο των πόλεων, όσον, αφορά την κάλυψη των κενών γνώσεων, γνώσεων για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σύνδεσμος που να συνδέει όλους κοινωνίες των πολιτών, κυβερνήσει, τα κτλ. σε ένα ισχυρό όχημα προς την πολιτική για την αλλαγή, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Μετά έχουμε και τη διασκέψη των πόλεων και των κλιματικών προσαρμογής που γίνεται κάθε άνοιξη όπου εκεί ακριβώς συζητάμε στα πλαίσια της ε, πολιτικής των προσαρμογών για το ρόλο της συγκεκριμένης κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρίσνικ, είχατε μια ερώτηση κύριε Μπρεσνικ. Ναι, ναι. Ε, πρέπει να απαντήσω τώρα όλες τις δύσκολε ερωτήσεις. Νομίζω ότι είχαμε έτσι ένα μείγμα ερωτήσεων για το πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των προγραμμάτων και των Ταμείων Συνοχής. Νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν στη διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού. Βέβαια, τα προγράμματα συνεργασίας είναι πιο εύκολα επειδή δεν έχουν τεράστια κονδύλια. Οπότε για μας δεν σημαίνει ότι χτίζουμε ας πούμε δρόμους ή χρηματοδοτούμε υποδομή κτλ. Οπότε το να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των προγραμμάτων μας για μας είναι πιο εύκολο γιατί είναι πιο εύκολο να πετύχει κανείς ισορροπίες στα πλαίσια των προγραμμάτων μας. Οπότε για μας το να μην χρηματοδοτήσουμε, ας πούμε, βιοκαύσιμα, ή με χρηματοδοτήσουμε βιοκαύσιμα ή αντίστοιχες δράσεις, για μας είναι πιο εύκολο. Ιδιαίτερα όσο περνάει ο χρόνος. Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 7-13 και την τωρινή και τη συμμετοχή στον πραγματισμό, νομίζω ότι η συμμετοχή εκεί μπορεί να βελτιωθεί. Οπότε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερο την άποψη των εμπλεκομένων σε σχέση με το τι θεωρούν αυτοί ότι είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και κατά πόσο θα μπορούσαμε να δώσουμε μια πιο ισχυρή φωνή στις πόλεις. Βέβαια η εμπειρία ποικίλει από χώρα σε χώρα σε σχέση με τη συμμετοχή. Και κατά πόσο επιτρέπεται ακριβώς τους εμπλεκόμενους να συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση προγραμματισμού. Πάντως, στο κανονισμό και στον σχεδιασμό των προγραμμάτων, αυτό που προβλεπόταν νομίζω ήταν θετικό, ώστε να ανοίξουν ακριβώ αυτά τα προγράμματα περισσότερο και να εμπλακούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι στην φάση του προγραμματισμού. Πάντως, νομίζω ότι είναι σημαντικό, μιας και υπάρχει ένας γεωγραφικός διαχωρισμός και βλέπουμε και τα σημερινά παραδείγματα, οι πιο προχωρημένοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγάλες, οι μεγαλύτερες πόλεις σε πλούσιες χώρες. Αλλά για να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να εμπλέξουμε και τις περιφέρειες που έχουν και, αυτοί, και αυτές προχωρήσει. Οπότε γι' αυτό τα προγράμματα πρέπει να είναι πιο εύκολα, να είναι πιο εύκολα στην πρόσβαση για αυτές τις ομάδες, δηλαδή ώστε και αυτές να, οι ομάδες ώστε και αυτές να συμμετάσχουν. Εγώ βρίσκομαι στη διαχείριση του τρίτου προγράμματος και βλέπω ότι υπάρχει μια καμπύλη μάθησης. Δηλαδή, έχουμε μια εξέλιξη. Αυτοί που απλά και μόνο ήταν αυτοί που συμμετείχαν παθητικά, τώρα έχουν ενεργητικό ρόλο. Έχουν λοιπόν καλύτερο ρόλο τώρα και προσπαθούν να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν. Αλλά βέβαια και ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να μειωθεί. Γιατί οι εταίροι των προγραμμάτων μόνοι τους δεν μπορούν ακριβώς να διεκπαιρεώσουν αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα γιατί υπάρχουν πολλές απαιτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλατε, κύριε Γκουαρντίνοβα, θα θέλατε να απαντήσετε κι εσείς. Πολύ σύντομα δύο σχόλια Οι πιο απομακρυσμένε περιοχέ αναφέρθηκαν. Να πω ότι είναι σημαντικέ βέβαια αυτέ και προετοιμάζουμε μία ανακοίνωση για φέτο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα χωριστά. Βέβαια και η κλιματική αλλαγή αφορά αυτές τις πιο απομακρυσμένε περιοχές. Να κάνουμε μια διευκρίνηση μόνο είχαμε το στόχο 20% για τις αζόρες, να απαντήσω στην ερώτηση στη σχετική, είχαμε το στόχο 20% στο ΠΔΠ. Είχαμε και τα κονδύλια για την οικονομία χαμηλό άνθρακα. Να σας παραπέμψω βεβαίως και στο μη περιφερειακή Ανάπτυξης που αφορά ακριβώς την οικονομία χαμηλό άνθρακα. Δεν ξέρω ακριβώ τι ισχύει τοπικά, αλλά βεβαίω μπορούμε να προβλέψουμε διαφορετικέ λύσει, όχι μόνο ενεργειακή απόδοση, αλλά ευφυή δίκτυα όσον αφορά τι ΑΠΕ, μεταφορέ, έρευνα και καινοτομία, καινοτόμε λύσει, ανάλογα ξαναλέω με τις ισχύουσε τοπικέ συνθήκε. Α πούμε θερμομόνωση ή μόνωση των κτηρίων μπορεί να είναι ε, ένα αποτελεσματικό μέτρο για την αντιμετώπιση του καύσωνα, όχι μόνο ας πούμε Τη ε, κλιματική αλλαγή, αλλά πιο συγκεκριμένα του καύσωνα. Κάπω έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να το δούμε. Ευχαριστώ. Και εγώ μια σύντομη παρατήρηση για την περίοδο μετά το 20 και το πι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Θα μπορούσαμε πούμε, να επιταχύνουμε τι δράσει που αφορούν την κλιματική αλλαγή σε σχέση με την περίοδο 14-20. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτό λέμε και με συνέχεια. Να μην ξεχνάμε την τωρινή περίοδο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις και τις συζητήσεις. Ευχαριστώ και πάλι. Συνεχίζουμε τώρα με την ημερήσια μας διάταξη. Κλείνουμε τη δημόσια συνεδρίασή μας και περνάμε στις συνεδρία των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ όσους δεν έχουν σχέση με τις συνεδρίες των συντονιστών να αποχωρήσουν.